I give the floor, uh, Mrs. Gill. Η κυρία Γκίλ έχει το λόγο. Uh, thank you. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ στήριξα αυτή την έκθεση και συγχαίρω την εισηγήτρια τα σκάνδαλα τα σχετικά του πρόσφατου παρελθόντος δείχνουν ξεκάθαρα το που μπορούν να οδηγήσουν ε, τα ανεξέλεγκτα αυτά μέτρα σύγκρισης καθώς χειραγωγούνται για να κλέψουν ε, τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Η Κομισιόν ε, επέβαλε ένα πρόστιμο 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπότε θα επηρεαστεί έτσι η καθημερινή ζωή των καταναλωτών καθώς με αυτά καθορίζεται το επίπεδο των τραπεζικών δανείων πάρα πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δε τράπεζες οι οποίες λένε ότι δεν έχουν λεφτά να δώσουν δάνεια, έδωσαν δισεκατομμύρια για τα πρόστιμα που έφαγαν. Οπότε η έκθεση είναι ισορροπημένη και αναλογική και νομίζω πως η διαφάνεια και η επίβλεψη της διαδικασίας αυξήθηκε και αντιμετωπίστηκαν ε, οι συγκρούσεις συμφερόντων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκίλ. Κυρία Πετήρ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η χειραγώγηση των ε, λεγόμενων πλαφών αυτών αναφοράς ε, μας δείχνει γιατί πρέπει ακριβώς να παρακολουθούμε την ε, χρήση τους. 400 δισεκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποιούνται σε μέσα χρηματοδότησης αποδεικνύουν πως η διαφάνεια στα δεδομένα και τις μεθόδους είναι πάρα πολύ σημαντική και έτσι θα λύσουμε το ζήτημα των συγκρόμενων συμφερόντων. Αυτά τα benchmarks χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί Παραδείγματο χάρη ε, το επιτόκιο, όπως είπαμε, στεγαστικών δανείων, κατά το οποίο προφανώς επηρεάζει αρνητικά τους καταναλωτές. Στην Κροατία είχαμε το σκάνδαλο των δανείων με ρήτρα ελβετικού φράγκου που οδήγησε πάρα πολλά νοικοκυριά στα όρια της καταστροφής. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Ο κύριος Φλάναγκαν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ε, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να ξέρουν ε, ε, για αυτά τα σκάνδαλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι πηγαίνουμε έτσι ώστε να μην αφήνουν τα λόμπι στα χνάρια τους πάνω σε όλα τα νομοθετήματα. Εν πάση περιπτώσει καλύτερα το λίγο από το τίποτα. Wolf. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, καταψηφίσαμε την πρόταση της ε, ε, Κομισιόν στην έκθεση της κυρίας Βανό Χούισεν όσον αφορά τους δείκτες αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα αυτά. Αυτοί οι δείκτες είναι πολύ σημαντικοί για τις συμβάσεις και μάλιστα υπάρχει ειδική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία καλύπτει τα θέματα αυτά. Εδώ χρησιμοποιούνται και άλλοι δείκτες για άλλα αγαθά και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε λιγότερους ε, δείκτες ε, με τον τρόπο αυτό ε, να δοθεί ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη γιατί φεύγουν θέσεις εργασίας από την Ευρώπη και επομένως έχουμε μικρότερη οικονομική ανάπτυξη επομένως εμείς θέλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι την Ευρώπη γιατί η Ευρώπη είναι αυτή η οποία διώχνει τις θέσεις εργασίας Ευχαριστώ πολύ. Τίτσο. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι πολύ σημαντική ε, αυτή η έκθεση και το νομοθέτημα για τους δείκτες στους χρηματοπιστωτικές συμβάσεις γιατί οδηγούνται σε κατακαιρματισμό οι αγορές ε, θεωρούμε ότι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενοποίηση αυτών των ε, αγορών. Ε, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με τα 17 ε, δις ευρώ που, ε, του προστίμου ε, για τον κακό χειρισμό των δικτών αναφορά το Δεκέμβριο του 2013. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά θέλουμε σωστούς δείκτες. Αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί έτσι ώστε να σταματήσουν ε, οι κακοί χειρισμοί όσον αφορά τους δείκτες αυτούς. Ε, συνεχίζουμε με την έκθεση ε, Πέδρο Σίλβα Περέρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Ο κύριος Χέις είναι ο πρώτος ομιλητής υπερψήφισα την έκθεση αυτή και συγχαίρω όσους συμμετείχαν στην έκθεση. Πρέπει να είναι σαφές ότι εμείς θέλουμε σοβαρά να επιτύχουμε τους στόχους, αλλά ε, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να σεβαστούμε και το 0,8%. Ε, υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες από, σιγά σιγά από την ύφεση πηγαίνουν προς την ανάπτυξη και τη προς την την ανάπτυξη και επομένως ε, θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Το δεύτερο σημείο ε, είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, να επιτύχουν ένα μεγαλύτερο μέρος του αναπτυξιακού προπολογισμού. Αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί να υπάρξει σημαντική ανάπτυξη, αλλά υπάρχουν περιοχές όπου α πούμε η Ποσαχάρη Αφρική αλλά και άλλε περιοχέ του κόσμου που υστερούν όσον αφορά την ανάπτυξη. Επομένω, θα πρέπει να αναπτυχθούν και οι περιοχές αυτές έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ. next uh, speaker is uh, Mrs. Gill. Η κυρία παρακαλώ. for development, because it is deeply disappointing that we are... Είναι πάρα πολύ απογοτευτικό ότι δεν έχουμε πετύχει τους στόχους χιλιετίας Πολλά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή δεν προσφέρουν το 0,7 του ΑΕΠ ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια. Πιστεύω λοιπόν πως έφτασε η ώρα τα κρατη να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Το κόστος ανθρώπινες ζωές, το κόστος... Το κόστος που αντιμετωπίζουμε με όσους εγκαταλείπουν την φτώχεια και τους πολέμους που δημιουργούν αυτή τη φτώχεια. Εάν λοιπόν τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη βρούμε μια ημερήσια διάταξη η οποία είναι πιο ε, σταθερή, θα πρέπει στην διάσκεψη της Αντισαμπέμπα ε, αυτό να μεταφραστεί σε μια πιο ισχυρή δέσμευση και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μιλήσουμε με μια φωνή ακολουθώντας την ίδια γραμμή. Χρειάζεται λοιπόν δράση για να βοηθήσουμε τα, υποανα... τα αναπτυσσόμενα κράτη να έχουν δικούς τους πόρους με πολιτικές που θα τους επιτρέψουν να σταθούν στα πόδια τους. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ολιμήτρια, η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ κόσμο που ακόμα ζει σε συνθήκες φτώχειας, που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία και κυρίως σε χώρες οι οποίες επηρεάζονται από σειράξεις, από σταθερότητα, από σταθεροποίηση, με συγχωρείτε. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Υπάρχουν οι πόροι στον πλανήτη έτσι ώστε σταδιακά να εξαλείψουμε αυτή την κατάσταση. Η έκθεση αυτή καλεί τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψουν το στόχο του 0,7% για την αναπτυξιακή βοήθεια. Πιστεύω όμως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική ε, διάσταση πριν βάλουμε κάποια όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Είναι μεγαλύτερη, ε, η μεγαλύτερη συνεισφορά η ευρωπαϊκή στον κόσμο ε, και καταλαβαίνετε πως οι πόροι που διαθέτουμε θα πρέπει να χρησιμοποιούν με το βέλτιστο δυνατόν τρόπο και δεν είναι κάτι που έχουμε πετύχει σήμερα. Η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να στηρίζει τι βασικέ κοινωνικέ υπηρεσίε και να δώσει δυνατότητε αυτοαπασχόληση σε εντόπιου πληθυσμού στην ε, γεωργία. Και νομίζω πω το τμήμα αυτό θα πρέπει να διαγραφεί από την παράγραφο 28 αυτή τη έκθεση. Επόμενο, η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστήριξα αυτή την έκθεση γιατί έχει πολύ σημαντικά κτήματα. Δηλαδή, οι χώρε με υψηλά εισοδήματα θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, χρηματοδότηση αναπτυαξή με πιο διαφορό τρόμα. Επίση, ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη. Και η έκθεση στηρίζει την αρχή τη ισότητα των φύλων, γιατί κομβικό σημείο θεωρείται αυτή για τι αναπτυξιακέ βοήθειε. Επενδύσει σε χώρου κομβικού. υγεία, παιδεία. Και έτσι η χρηματοδότηση ερώτηση αυτή να λαμβάνει πάντα υπόψη το πώς, πώς ζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια. Ξέρετε πως στηρίζουμε την αναπαραγωγική ε, υγεία και τα δικαιώματα. Θυμόσαστε το δημοψήφισμα για τις αμβλώσεις στην Ιρλανδία. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να στηριχθούν αυτά όπως και τα υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δίνω το, ρόλο, το, το λόγο τώρα στην κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς πρέπει να αλλάξει η κατάσταση όταν μιλάμε για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, ζητήματα διαφθοράς ε, που προωθούν αυτό το φαινόμενο και θεωρώ πως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά στην πηγή τους. Τα τεράστια κέρδη λοιπόν που υπάρχουν ε, σε διάφορους ε, παράγοντες ε, ακριβώς επιδεινώνουν την κατάσταση αυτή ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από διάφορες περιοχές και των ανθρώπων που τους εκμεταλλεύονται. Και αποτελεσματικές λύσεις ανάπτυξης ε, και η αντιμετώπιση της διαφθοράς ε, και των φορολογικών παραδείσων είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη έκθεση για την παροχή υγείας στην Ευρώπη. Ρόντε έχει το λόγο. Mr. Κύριε Ρόντε. Ευχαριστώ πολύ. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε στην Ευρώπη είναι να διασφαλίσουμε ε, ότι θα έχουμε περισσότερες, ε, περισσότερους επιχειρηματίες και ότι ε, θα έχουμε καλύτερη εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εράσμους που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους νέους επιχειρηματίες ε, το σημαντικό βέβαια είναι ε, να ε, έχουν τα κράτη-μέλη ένα τέτοιο σύστημα στήριξης των, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας πρωτοβουλειών. Θα πρέπει να σταματήσουμε πια, να, να βγάλουμε από πάνω μας τα νομοθετήματα τα οποία είναι πλεονάζοντα και μη αποτελεσματικά. Θα πρέπει κράτη-μέλη να ε, έχουν ίσους όρους ε, έτσι ώστε να μπορούν ε, οι νέοι να ξεκινήσουν. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ιγκλέσια. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς υπερψηφίσαμε την έκθεση αυτή για πιο ασφαλή πρόσβαση στην υγεία στην Ευρώπη για να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις περικοπές και να εξασφαλίσουμε πως θα υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες στον κλάδο. Επιτρέψτε μου να σας επιστήσω την ε, προσοχή στο τι συμβαίνει με την υγεία στη χώρα μου, που ήταν ένα από τα συστήματα υγεία από τα πιο αποτελεσματικά στον κόσμο μέχρι πρόσφατα. Οι πολιτικές που ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα στην χώρα μου έχει καταρακώσει το κλάδο τη υγεία μέσω τη ιδιωτικοποίηση ε, και βεβαίω λόγω περικοπών. Μία χειροτέρευση πολύ επιθετική σε περιοχέ όπω η Βαλένσια ή η Μαδρίτη. Να σας υπενθυμίσω πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βασίστηκε στην ιδέα τη της δημοκρατίας που βασίζεται σε κοινωνικά δικαιώματα και σε κοινωνικές υπηρεσίες. Η χειροτέρευση της υπηρεσίας υγείας δεν χειροτερεύει μόνο την δημοκρατία αλλά και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ε, πλήττεται ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκίλ, έχετε το λόγο. Εγώ στήριξα την έκθεση για το θέμα αυτό, για την ασφαλεία στη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη. 10% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία πλήττονται από κάποιο είδους ατυχές γεγονός όσο βρίσκονται στο νοσοκομείο. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή 4,1 εκατομμύριο πολίτες μας ε, υποφέρουν από ασθένεια που ε, στοιχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν. Μεγάλο το κόστος. Το καλό είναι ότι μπορούμε αυτές τις ασθένειες σε μεγάλο ποσοστό να τις αποφύγουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας βοηθήσει να το πετύχουμε το να ελαφρύνουμε το βάρος που αντιμετωπίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας, τα οποία ήδη ασθενούν σε αρκετά κράτη ε, μέλη και ε, βεβαίως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημαίνει πως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ε, την χρήση νέων αντιβιωτικών και να ρυθμίσει τη χρήση αυτών. Και βεβαίως να δούμε πως οι ασθένειες δεν σταματούν στα σύνορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να πετύχει αποτελέσματα που ένα κράτος μέλος μόνος του δεν μπορεί να πετύχει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει το θέμα αυτό να αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε καλύτερη επιτήρηση, καλύτερη συλλογή ε, δεδομένων για τις ασθένειες που σχετίζονται με ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ρόπε. Έχετε το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος πως η έκθεση αυτή είναι από τις σημαντικότερες εκθέσεις ε, στην θητεία αυτή. Αυξάνεται η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά δεν είναι κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει η προληπτική χρήση τους ε, στην ε, κτηνοτροφία. Όλο και περισσότερα ζώα πλέον ε, έχουν μικρόβια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα αντιβιωτικά και υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθούν στα τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους αγρότες και να έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες και για την παροχή αντιβιωτικών στους ανθρώπους. Το 2009, λόγω της γρήπης των χείρων, άρχισε ο κόσμος να αγοράζει αντιβιωτικά στην ε, Λιθουανία, αλλά χρειάζονται και πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες στη συσκευασία. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Πέτυρε, τα συστήματα υγείας πάντα πλήττονται από τα μέτρα λιτότητας, ε, πάντα κατόπιν συμβουλών διεθνών οργανισμών. Εγώ είμαι υπέρ ενός συστήματος στα λειτουργία, αλλά όχι υπέρ των περικοπών. Γι' αυτό στήριξα αυτή την έκθεση. Η Κομισιόν το 2012 είδε πως η ασφάλεια των ασθενών ε, κινδυνεύει άμεσα από τα μέτρα λιτότητας και τις περικοπές στην υγεία που επηρεάζουν άμεσα την παροχή υγείας. 8-12% των ασθενών ε, πλήττονται κατά τη διάρκεια της νοσηλεία τους. 30% αυτών των περιπτώσεων είναι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Ε, Παραδείγματο χάρη το να δίνουμε φάρμακα που δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρωση, κατάχρηση των αντιβιωτικών. Μαζί με τις άλλες ε, συνέπειες της ε, της χρήσης φαρμάκων οδηγούν σε ένα κόστος 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πέδρε, υπερψήφισα την έκθεση για ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη, διότι είναι πλήρης και επαρκής. Ταυτόχρονα θέλω να καταγγείλω ότι στην Ελλάδα, 7 χρόνια μετά την επιβολή του ΆΜΚΑ, του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με το νόμο 3655-2008, εκατοντάδες χιλιάδες έλληνες πολίτες στερούνται παράνομα κάθε υγειονομική περίθαλψη τα κοινωνικά επιδόματα και τις συντάξεις επειδή για λόγους θρησκευτικής συνείδησης και προστασίας των συνταγματικών τους ελευθεριών αρνούνται να λάβουν άμκα. επειδή λοιπόν αρνούνται την περαιτέρω αριθμοποίηση του ανθρώπινου προσώπου τιμωρούνται και αποκλείονται από το σύστημα υγείας έτσι πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους φάρμακα εξετάσεις χειρουργικές επεμβάσεις ακόμη και αν έχουν καταβάλει κανονικά τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. πρόκειται για ένα κοινωνικό ρατσισμό που πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα και για τον λόγο αυτό θα εντείνω τον αγώνα μου και εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Νέκοφ. Επομένως, έχουμε τον κύριο Κέλλη, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Χθες ε, στο βράδυ είχαμε την συζήτηση για το θέμα αυτό και ε, χαίρομαι γιατί είχα την ευκαιρία να ακούσω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ε, και μίλησα και όλα στη διάρκεια αυτής της συζητήσεως. Εμείς ψηφίσαμε ε, ε, κατά μεγάλη πλειοψηφία 637 ψήφοι υπέρ με 679 ψήφους ε, επί 679 ψηφισάντων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό βεβαίως να μπορούμε να θεραπεύσουμε τους ανθρώπους αλλά κυρίως θα πρέπει προληπτικά να τους προστατεύσουμε έτσι ώστε να μην αρρωστήσουν, να προβλέπονται φυσικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, να προβλεφθούν οι απαραίτητες έκτες υποδομές ε, που θα δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο να περπατάει, να κάνει jogging, ε, να κάνει ποδήλατο ή να πηγαίνει στην πισίνα και έτσι η πρόληψη θα είναι ε, καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάρκιν, τελευταία ομιλήτρια του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ στήριξα την τροπολογία που ζητάει από την Κομισιόνα νομοθετικό πλαίσιο για τα νέα αντιβιωτικά οι 27.000 ε, ε, ε, είναι αυτοί 25.000 πέθαναν από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και ελλειπή αντίσταση στα αντιβιωτικά στην χώρα μου σε ένα χρόνο. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Ο δόκτωρ Τόνι Χόλαντ από το Υπουργείο Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται άμεση βοήθεια και δράση γιατί μπαίνουμε σε μια χρονική περίοδο όπου ακόμα και ελάσσονο σημασία ιώσεις ή λοιμώξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν το θάνατο του ασθενού ε, στην ε, ε, Ιρλανδία δύο φορές περισσότερο χρησιμοποιούνται οι θεραπείες ε, με αντιβιωτικά και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της υπερσυνταγογράφησης αντιβιωτικών κυρίως στους ηλικιωμένους της Ιρλανδίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε για αυτή την υπερσυνταγογράφηση να ληφθούν άμεσα μέτρα γιατί ο συνολικός πληθυσμός αλλά και οι ηλικιωμένοι κυρίως τίθενται σε μεγάλο κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκιν και περνάμε στην επόμενη επόμενη έκθεση είναι η έκθεση DeBacker ε, όσον αφορά τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης στις τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτος ε, ο μιλητής, ο κύριος Ρόντε. Κύριε Ρόντε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπέρδεψα τα πράγματα. Γιατί αυτά που θα πω τώρα, αυτά που είπα πριν ήταν αυτά που ήθελα ε, να τα πω τώρα. Μίλησα για την επιχειρηματικότητα, ενώ το θέμα μας προηγουμένως ήταν η υγεία. Ε, ε εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι πολλοί εκτός από τους διερμηνείς κατάλαβαν ότι μιλούσα για λάθος ε, θέμα. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως... Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επαναλάβω αυτά που είπα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως που μου δώσατε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Ρόντε. Δεν βλέπω την κυρία Μολινάρ. Next speaker is, uh, Mr. Balzo. Ο κύριος Μπαλτζό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ε, στηρίξαμε την έκθεση αυτή γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην πράσινη οικονομία. Υπάρχει μεγάλη αγορά, ένα 3 εκατομμύριο ευρώ ετησίως ε, και μπορεί το 2020 να έχει διπλασιαστεί. Γιατί πρέπει λοιπόν να εμπλακούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός. Πρέπει να θυμάμαστε ότι 67% των θέσεων εργασίας στην Ένωση δημιουργούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να εμπλακούν στην υπόθεση αυτή, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε κονδύλια και πρέπει να πω πως το βρίσκω κάπως περίεργο πως όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών Επενδύσεων τα πλεονεκτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε ωφελούν επιχειρήσεις από, με 3.000 υπαλλήλους, δηλαδή όχι τόσο μικρομεσαίες. Ευχαριστώ. κυρία Νίνα Γκίλ. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο σημαντικό να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης μόνο, αλλά να μειωθεί και το κόστος του πρασινίσματος στην περιοχή μου τα δυτικά Midlands ε, η χρηματοδότηση της Ένωσης ε, έχει δοκιμήσει, ε, έχει οδηγήσει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα τέτοιων υπηρεσιών, ίσως τον μεγαλύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου δε του ότι, ότι οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρειά μου λένε πως δεν βρίσκουν ακόμα τέτοια χρηματοδότηση πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Αλλά εγώ το υπερψήφισα και για τους λόγους που ανέφερε η ομάδα μου. Ότι δηλαδή θα δώσουμε την σωστή προσοχή στις μικροεπιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούμε πλήρως την δυνατότητα που έχουν για να υπάρχει και συνέργεια και επιχειρηματική πόλη. Έτσι θεωρώ πως χάσαμε μια ευκαιρία γιατί δεν γίνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ πολύ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την ανάγκη κάποιας νέας όθησης για την ανάπτυξη και για να διατηρήσει η Ευρώπη τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα τα οποία ήδη ε, έχει ή απολαμβάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειήσει το κόστος όπως επίσης ε, και τις δαπάνες για εισαγωγές για παράδειγμα ενέργειας. Έχουμε λοιπόν την πράσινη οικονομία που θα μπορούσε με τη συμμετοχή του ιδιωτικού κλάδου να μας κατευθύνει προς την σωστή ε, κατεύθυνση. Δεν μπορούμε όμως να το θεωρούμε ως αυτόνομο στόχο. Η οικονομική θέση της Ευρώπης θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη ε, κατάσταση για τους πολίτες μας. Και τα στοιχεία που έχουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας οδηγούν στο εξή συμπέρασμα. Το 89% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ε, μικρομεσαίες. 67% των θέσεων εργασίας προέρχονται από αυτός και είναι το 50% της προστιθέμενης αξίας στην εργασία. Αυτές λοιπόν να μας οδηγήσουν και να μας κατευθύνουν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέει ο κύριος Μπέντσεν, έχω στηρίξει αυτή την έκθεση. Είναι πολύ καλή πρωτοβουλία και θα δώσει πλεονεκτήματα στην Ευρώπη. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την διαβάσει έτσι ώστε αυτές οι πρωτοβουλίες να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δυναμικό που δεν χρησιμοποιείται, που μπορεί να μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς, να κάνει πιο ανταγωνιστικές εταιρείες μας στις υπηρεσίες και στις κλάδους παραγωγής. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο ρυθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πολύ ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά και θα μπορούσαν να προσφέρουν λύσεις. Λύσεις για προϊόντα, όπως επίσης και για πράσινες υπηρεσίες, όπως ε, η διαχείριση εγκαταστάσεων, η συντήρηση εγκαταστάσεων. Αυτό είναι σημαντικό. Μιλάμε για τις πράσινες υπηρεσίες που θα δώσουν πωλήσει, που θα δώσουν κέρδος και αυτά μπορούν να ενταχθούν και σε μελλοντικές ε, εμπορικές συμφωνίες, όχι μόνο στην TTIP. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν βλέπω τον κύριο Νεκόφ. Next speaker uh, Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χάναν. Κύριε Χάναν. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπει κανείς τι κρύβεται πίσω από τα πράγματα. Γιατί μιλάμε για πράσινες πολιτικές. Εάν θέλετε να πείτε κοστίζει. Κοστίζουν οι οικολογικοί στόχοι. Χρειαζόμαστε για να μην υπάρχει υπερθέρμα στο πλανήτη να έχουμε χαμηλότερα κέρδη. Εντάξει, πείτε το έτσι, απερίφραστα είναι πιο ειλικρινέ. Αλλά το να πείτε πω με τρόπο αυτό θα προωθήσετε την οικονομία αποτελεί τέτοιου είδου μη αποδεδειγμένη οικονομική ε, υπόθεση που είναι σαν να μας λέτε πως αν προσλάβει περισσότερους η κυβέρνηση θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θα πληρώνουμε περισσότερους φόρους και θα αναπτυχθεί η οικονομία. Μα στη Σοβιετική οικονομία ε, κάναν κάτι τέτοιο και είδαμε που οδηγήθηκαν. Έχουμε λοιπόν τη θεωρία των εμφανών και αφανών ε, κοστών. Ε, είναι αυτή η οικονομική θεωρία που λέμε πως οι θέσεις αυτές της εργασίας όσο κοστίζουν τόσο πολύ να δημιουργηθούν που δεν θα δώσουν κάτι στην οικονομία. Δεν είναι οι πράσινες πολιτικές που δημιουργούν ανάπτυξη, είναι η ανάπτυξη που δημιουργεί πράσινη πολιτική. Γιατί ε, με τον τρόπο αυτό προσφέρει... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χάναν, έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Ο κύριος Κέλλη. Καλημέρα σας. Θα ήθελα κι εγώ να σας πω πως χτες το βράδυ που το συζητήσαμε Ακούσαμε τα όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πραγματικά περιέγραψε ποιες είναι οι συστάσεις της έκθεσης και η πλειοψηφία εδώ μας είπαν πως είναι υπέρ. 519 υπερψηφίσαμε από τους 672 που ψήφισαν. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχουν τέτοιου είδου ευκαιρίες που θα πρέπει να δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν ένα ε, συστατικό πολύ σημαντικό της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας, 87% ε, των εταιριών και τα λοιπά, το 67% των θέσεων εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν το, η τέτοιου είδους σκέψη που ότι πιο μικρός θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο κτλ θα είναι πολύ επιβοηθητικέ και θα πρέπει να ε, ξεπεράσουν και τις γραφειοκρατίες οι οποίε είναι μεγαλύτερη απειλή για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πρόσβαση στις πιστώσεις. Αν τα καταφέρουμε αυτά όλα νομίζω πως θα πετύχουν και οι πολιτικέ μα για τι μικρομεσαίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Εγώ στήριξα αυτή την έκθεση και ειδικά την τροπολογία εκείνη που ζητάει από την Κομισιόν να αποσύρει παροχημένη νομοθεσία. Με απλά λόγια να κόψει την, ε, να μειώσει τη γραφειοκρατία. Πάντα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικής και αναλογικής ε, ρυθμισής. Ε, και σε πολλές περιπτώσεις εδώ πέρα επιβάλλουμε βάρη τα οποία δεν πετυχαίνουν καν τους στόχους τους ξανά και ξανά ακούμε τους πολιτικούς να παραπονιούνται για τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Και συνήθως βεβαίω κατηγορούν τις Βρυξέλλες. Όταν όμως έχουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν για να καταργηθεί γραφειοκρατική και παροχημένη νομοθεσία, πολλοί την καταψηφίζουν. Ε, δεν γίνονται όλα, ή το ένα ή το άλλο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαλετίτς τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για τις δυνατότητες της πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών και τονίζει την ανάγκη σωστής ε, πληροφόρησης ε, για τους επιχειρηματίες. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια της Ένωσης για να επιτευχθεί μια μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας προωθούν την ανάπτυξη και πρέπει να τις βοηθήσουμε για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στήριξα την έκθεση The Backer, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να υπάρξει πράσινη ανάπτυξη, για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Ε, Ευχαριστώ.